μερίσες διάταξη στην έκθεση της κυρίας Μπόουλς με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών. Το λόγο έχει καταρχήν η εισηγήτρια η κυρία Μπόουλς. Παρακαλώ. National and regional account. Οι εθνικοί και περιφερειακοί λογαριασμοί είναι ο κρογωνιαίο λήθο όλων των μακροοικονομικών στατιστικών και είναι το πρίσμα από το οποίο εξετάζουμε τι οικονομίε μα. Όλοι συμφωνούμε ότι ε, θα πρέπει να έχουμε σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ισοτική σημασία. Σκεφτείτε την έναρξη τη ε, οικονομική κρίση, χειραγώγηση στατιστικών στοιχείων, η παροχή ανακριβών πληροφοριών. Έχουν ολέθρια αποτελέσματα ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ήταν μακροχρόνιος στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η βελτίωση των στατιστικών στοιχείων και η αύξηση των αρμοδιοτήτων της Eurostat. Η Eurostat όμως ε, εξαρτάται από την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνει. Κάναμε πολλά στο εξαπλό και το διπλό πακέτο για να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Στο δημοσιονομικό πλαίσιο του εξαπλού πακέτου συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνεται καλύτερη αναφορά των ε, ε, δημοσίων ε, οικονομικών και των δημοσίων δαπανών. Αλλά χρειαζόμαστε και ακριβείς στατιστικές πληροφορίες. το 2010 έχουμε ένα κανονισμό με δύο παραρτήματα. Το ένα αφορά κατάλογο ε, στοιχείων που θα πρέπει να συλλέγονται και που είναι αυτονόητος ε, ε, και το παρέρτημα Α περιλαμβάνει στατιστικές και λογιστικές μεθοδολογίες. Είναι εκατοντάδες σελίδες και οι γλωσσομαθείς νομικοί της γραμματείας το έλεγξαν και μου επισήμαναν πολλά ενδιαφέροντα σημεία και τους ευχαριστώ θερμά. Ε, με τις διαδοχές μεταρρυθμίσεις, ε, οι δαπάνες ε, και η και τεχνολογική ανάπτυξη μετατράπηκε σε δημιουργία κεφαλαίου που αντανακλά την οικονομική κατάσταση, κάτι που επηρεάζει το ΑΕΠ και την κατανομή των διαρθρωτικών κονδυλίων. Αυτό όμω θα φανεί περισσότερο μέχρι το 2020 και ο αντίκτυπο είναι μικρός. Θα πρέπει να ελέγξουμε και την πορεία του χρέους. Στι τριμερείς διαλόγους η διαπραγματευτική εντολή τη αντιπροσωπεία μας ήταν σαφή. Θέλουμε ποιοτικέ στατιστικές, πληροφορίες, διαφάνεια και όσο το δυνατόν λιγότερες παρεκκλήσει από τι υποχρεώσει των κρατών μελών. Κάποιε μικρέ χώρε έχουν κάποιες ευνόητους λόγους ε, για το ότι δεν παρέχουν το ίδιο αριθμό στατιστικών πληροφοριών στη Eurostat όπως οι μεγάλες χώρες, αλλά θα θέλαμε οι εξαιρέσεις να περιοριστούν στο απολύτως απαραίτητο, να γίνεται τακτική αναθεώρησή τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθά ε, μεθοδολογικά τα κράτη-μέλη όταν το ζητήσουν, προκειμένου να σταματήσουν ενδεχομένω οι παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις και νομίζω ότι με τη διατύπωση το πετυχαίνουμε κάτι τέτοιο. Το πιο ακαθόδε σημείο ήταν ε, όταν τέσσερις μεγάλες χώρες ε, μέλη κατάχθηκαν ε, κατά της ε, υποχρεωτικής διαβίβασης των ε, πληροφοριών για τις υποχρεώσεις καταβολής συντάξεων, όπως προβλέπει η οδηγία για το εξαπλοπακέτο. Κάτι που είναι παράδεκτο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ε, κατάφορη προσπάθεια να κρατηθούν ευαίσθητες πληροφορίες κρυφές και να μην εντάσσονται στους υπολογισμούς. Και μάλιστα προβάλαμε αυτό το σημείο στον τύπο και διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος είναι με το πλευρό μας. Θέλουμε τώρα μια έντιμη συζήτηση για τους δημόσιους λογαριασμούς. Αν, επιτρέψουν, αν επιμένουν τα κράτη-μέλη να κρύβουν κάποιες ε, άβολες ε, και σκληρέ αλήθειε. Τελικά με τι διαπραγματεύσει καταλήξαμε συμφωνία ότι όλα τα κράτη-μέλη θα μεταβιβάζουν τα σχετικά στοιχεία, θα διαβάζουν τα σχετικά στοιχεία και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια. Έχουμε και άλλα επιτέγματα στην έκθεση και ευχαριστώ θερμά του και οδησηγητέ για τη συνεργασία του, ε, γιατί πολλοί θεώρησαν το θέμα αυτό σχετικά ενιαρό, αλλά είχε και κάποια συναρπαστικά σημεία όπως σας είπα και επίσης θα αποτελέσει θεμελιώδες εργαλείο για τη σωστή και χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ κυρία Μπόλς. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Ποτότσνικ για να μας παρουσιάσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχω την τιμή να σας απευθύνω εξ ονόματος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα του συναδέλφου Αλγίντα Σέμετα που είναι αρμόδιο για το χορτοφυλάκι αυτό. Ε, ποιος είναι ο στόχο του κανονισμού που προτείνεται είναι η αναθεώρηση, ενημέρωση και βελτίωση ε, του σημερινού συστήματος ε, S95 για τους λογαριασμούς στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών που πρόσφατα ενημερώθηκε για να είναι τα στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα και ενημερωμένα. Είναι μεγάλο εγχείρημα, ε, έτσι ε, θα ε, τεθούν τα θεμέλια για τους εθνικούς λογαριασμούς για πολλά χρόνια. Για μας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών για τους ιδίους πόρους, για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, για τα διευθυντικά ταμεία και για την ανάλυση του συντονισμού και της σύγκλησης των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Η αναθεώρηση του συστήματος ΕΣΑ βασίστηκε σε ευρεία διαβούλευση των εθνικών εμπειρογνωμόνων, των χρηστών και ε, των ε, ε, όσων παράγουν και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη. Είναι καλά σταθμισμένο ως προς τις ανάγκες των χρηστών σε δεδομένα και ως προς το φόρτο που υφίστανται οι διοικήσεις. Ε, μετά από τριμερή διάλογο ε, συμφωνήθηκε ένα συμβαστικό κείμενο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, με στόχο να συμφωνηθεί σε πρώτη ανάγνωση η πρόταση. Εμείς υποστηρίζουμε στεναρά το συμβαστικό κείμενο γιατί έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει τα απαιτούμενα δεδομένα για τις πολιτικές της και να ασκεί και τον ελεγκτικό της ρόλο. Ακόμα και αν Υπάρχουν κάποια στοιχεία που αποκλίνουν από την κοινή αντίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για τις κατεξουδότητε πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι το άρθρο 290 της συνθήκης θα πρέπει να ερμηνευτεί ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτόνομη στην προετοιμασία των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Η συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων αντανακλά την ερμηνεία αυτή του παρόντος άρθρου. Γιατί ε, ε, απέρχεται από αυτή την ε, συμφωνία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μπόλς, για τη βαθιά της προσήλωση και στους στόχους και χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων πιστεύω ότι φτάσαμε στον κοινό μας στόχο για ένα πολύ γερό σύστημα πλαίσιο εναρμόνισης των στοιχείων, των στατιστικών στοιχείων ε, των εθνικών, έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς και οι κυβερνήσεις να βασίζουν τις αποφάσεις τους. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί ε, στην υλοποίηση θα ελέγχει την πλήρη εφαρμογή και από τα κράτη-μέλη του νέου συμφωνηθέντος πλαισίου έτσι ώστε τα στατιστικά στοιχεία που μας χρειάζονται να είναι πραγματικά στη διάθεσή μας και θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που αναλάβαμε απέναντι στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης προσβλέπει πάρα πολύ στη συνέχιση ενός γόνιμου διαλόγου με ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή που είναι εκ των όνων για να έχουμε στοιχεία υψηλής ποιότητας, αξιόπιστα, όσο και εθνικούς λογαριασμούς και άλλες μακροοικονομικές στατιστικές για να είναι υγιής η πολιτική που ασκείται και υιοθετείται γενικότερα προς όφελος της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για ένα λεπτό έχει το λόγο κύριε Χούμπνερ. Για πολλά χρόνια δεν υπήρξε πρόοδο στο σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών σε ό,τι αφορά το περιφερειακό επίπεδο, ενώ έχει αυξηθεί η ευθύνη του προϋπολογισμού των περιφερειακών ε, διοικήσεων και ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού των κρατών μελών που ξεπερνάει σε ορισμένα κράτη το 50% το διαχειρίζονται οι περιφερειακές αρχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανεί τα στοιχεία των περιφερειακών αρχών για να κατανοεί τις ε, εθνικές, τους εθνικούς λογαριασμούς, να καταλαβαίνει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, να καταλαβαίνει τη συμπληρωματικότητα διαφόρων παρεμβάσεων χρηματοδότησης για να βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητα των επενδύσεων και της χρήσης των πόρων και επίσης να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, ιδίως στον τομέα της, ε, της Η συμπίληση και αναφορά στοιχείων θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να γνωρίσουν καλύτερα το σχήμα των δαπανών σε περιφερειακό επίπεδο και την πραγματική ε, αποτελεσματικότητα και τον αντικτύπο αυτών των δαπανών. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε τώρα στους ομιλητές οι οποίοι λαμβάνουν το λόγο εξωρωματός των πολιτικών ομάδων τους. Πρώτος εκ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για δύο λεπτά ο κύριος Στόλογιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα. Θέλω να ευχαριστήσω κυρία Μπάουλς για το θαυμάσιο έργο της που αντανακλάται σε αυτή την έκθεση. Όλοι ξέρουμε τι προβλήματα έχουμε με τα μακροοικονομικά στοιχεία που έχουν δώσει ορισμένα κρατημέλη, στρεβλωμένα εθνικά ελλείμματα, έλλειψη κανόνων και έλλειψη κανόνων για να αναφέρουν τις δυνητικές χρεώσεις και τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε πιο εναρμονισμένους καραλινώνες με μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους κύριους εταίρους μας σε εμπορικό επίπεδο. Είναι το τελικό σημείο απόλυξη μια μακρά πορεία η έκθεση τη κυρία Μπάουλ και αυτό ανταποκρίνεται στι δικέ μα αιτήσει. Γι' αυτό η πολιτική μου ομάδα θα υποστηρίξει αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ τα μάλα. Ευχαριστούμε κύριε Στόλογιαν. Εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, για δύο λεπτά ο κύριος Σάντσεφ Πρεσέδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από το έργο της κυρίας Σάρων Μπάουλς και των σκιωδών εισηγητών, κυρίως του κυρίου Τσικλούνα, τον οποίο εγώ αντικαθιστώ και θέλω να τον ε, συγχαρώ για την εκλογή του στο Κοινοβούλιο της Μάλτας. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι στατιστικές είναι κεφαλαιώδεις για τη λειτουργία της οικονομίας και της δημοκρατίας βελτιώνουν τις γνώσεις των οικονομικών εταίρων και την οικονομική διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε στατιστικές ποιότητες, οι οποίες δίνουν στοιχεία ανεξάρτητα, αμερόληπτα, συγκρίσιμα, αξιόπιστα και έγκαιρα. Και να υπάρχει βέβαια τακτικός τρόπος με τον οποίο διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές. Το σύστημα τοπικών, περιφερειακών και εθνικών λογαριασμών ανέρχεται στο 1970 και βασίζεται σε ένα κανονισμό του 1976 δημιουργήθηκε επί τη βάση του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών. Η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου που έχουμε ενώπιόν μας προσαρμόζει το σύστημα αυτό στο σύστημα που προτείνει η Επιτροπή Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών από το 2009. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε την διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Οι τροπολογίες αυτές έχουν σαν στόχο να έχουν πληρέστερα στοιχεία, τονίζοντα πάντα την ανάγκη τη εμπιστευτικότητα και τη καλύτερη μεθοδολογία για θέματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό τομέα, το περιβάλλον, την έρευνα και την ανάπτυξη. Επίση, προωθούν μια καλύτερη κοινή ονοματολογία για τα περιφερειακά στοιχεία τη πολιτική συνοχή, ενισχύουν την οικονομική ε, σχέση μεταξύ των διαφόρων τομέων και εξασφαλίζουν μεγαλύτερο συντονισμό και βιωσιμότητα στις συντάξεις. Επομένω, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες χαίρονται για τη συμφωνία αυτή η οποία επιτεύχθη σε επίπεδο πρώτη ανάγνωση και ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ε, από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, Αντολίνε. Εκ μέρου τώρα των φιλελευθέρων, για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Τρεμόσα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή είναι σημαντική γιατί είναι από τις λίγες εκθέσεις όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει ε, και έχει λάβει υπόψη τη σημασία του περιφερειακού επίπεδου, της περιφερειακής διάστασης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναμειχθεί πιο ενεργά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις στατιστικές των περιφερειών για να διαμορφώσει μια σαφέστερη εικόνα για το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, δεν έχουμε διαφάνεια και οι πολίτες ε, δεν γνωρίζουν την εδαφική κατανομή των δημοσίων δαπανών της Ισπανικής Κεντρικής Κυβέρνησης. Επίσης, άγνωστοι είναι για τους πολίτες η σύλλογη των φόρων σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί εξασφαλίζεται σε κεντρικό μόνο επίπεδο. Αυτή η αδιαφάνεια της κεντρικής κυβέρνησης είναι ένας από τους λόγους της έξαρσης της των τάσεων στην Καταλωνία. Επίσης ε, θα πρέπει να αναλύσουμε την ε, αλληλεξάρτηση των ε, κρατών με τις περιφέρειές τους. Γι' αυτό οι φιλελεύθεροι θα υποστηρίξουν την έκθεση της κυρίας Μπόλς και θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε θερμά για, για την πολύ αξιόλογη προσπάθειά τους. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Το λόγο έχει εκ μέρους των Πρασίνων ο κύριος Φεν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι ελπιδοφόρο και χαρμόσυνο ότι βελτιώνονται οι κανόνες για τους εθνικούς κανονισμούς με δείκτες κοινωνικούς και οικολογικούς και είναι τα στατιστικά στοιχεία πλέον καλύτερης ποιότητας. Δεν θα πρέπει όμως να αποκρύψουμε ε, τι καθυστέρησε μήνες ε, αυτή την υπόθεση. Υπήρξε πολύ σκληρή αντιπαράθεση με κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο που δεν ήθελαν διαφάνεια ακριβώς ε, στον τομέα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσει. Ιδιαίτερα στην επιβάρηση των ε, ε, συντάξεων αλλά και αλλού στις δίτα, ας πούμε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που είναι εκτός ε, ισολογισμών. Είναι κρίμα γιατί κληθήκαμε να καλύψουμε το κόστος της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης και βλέπουμε ότι τα κράτη παραμένουν απρόθυμα να έχουν διαφανή προσέγγιση. Παραμένει ε, ελκυστικό να χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις από συγκάλυψη των κινδύνων και των εξόδων ε, αντί να προσελκύονται με σωστό τρόπο. Και είναι ακριβώς κρίμα που η Γερμανία ε, που ε, είναι υπέρ της τάξης και της πειθαρχία τώρα βρίσκεται ε, σε λάθος μεριά. Τι σημαίνει θα πάμε στον επόμενο γύρο της αντιπαράθεσης αλλά κάποια στιγμή θα υποχρεωθούν και οι χώρες όπως και οι επιχειρήσεις να έχουν κανόνες όπου υπάρχουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα τα δούμε αυτά τέλη του έτους θα τα ξαναπούμε και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Βίκη Φόρτ. Ευχαριστώ. Οι κυβερνήσεις ε, και οι δημόσιοι οργανισμοί ε, συλλέγουν χρήματα από τους φορολογούμενους, οπότε είναι εύλογο να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι που πηγαίνουν τα χρήματά τους ε, και τι έχουν, ποια είναι τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των κυβερνήσεων. Ε, ασχολήθηκα με το εξαπλό πακέτο και 27 χώρες ε, μέλη συμφώνησαν ε, να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους, τον ισολογισμό τους και τον εθνικό λογαριασμό τους. Βέβαια τώρα ως προς λεπτομέρειες ε, μερικές χώρες ε, ε, υπαναχωρούν και λένε ότι διαφωνούμε και δεν θέλουμε υποχρεωτικά να διαβάζουμε τέτοια στοιχεία. Οι μικρές χώρες είναι που τους επανέφεραν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και λένε στο όνομα των φορολογουμένων και για χάρη τους θα πρέπει να δημοσιεύεται τον τρόπο που χρησιμοποιείται τα δημόσια κονδύλια. Και ευχαριστώ θερμά τις μικρές ομάδες που ύψωσαν το ανάστημά τους υπέρ της διαφάνειας και υπέρ των των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων και περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Πρώτα για ένα 1,5 λεπτό. Το λόγο κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και ε, την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Μεταξύ άλλων, διότι Ε, σε όλες τις εκθέσεις που ασχολούνται με στατιστικές έχω πει επανελειμμένα ότι πρόκειται για στοιχεία, δεδομένα, αριθμούς που θα πρέπει να είναι πάντα ακριβή, συγκρίσιμα και αξιόπιστα. Να προέρχονται από συγκρίσιμες πηγές και να εντάσσονται σε ένα γενικότερο σύστημα για να μπορούν να αξιοποιούνται. δεν είναι άνευ ε, σε ποια στοιχεία βασίζονται οι αναλύσεις μας. Καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, υπερβολικά, είτε οποιημένα είτε υπερβολικά αρνητικά. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό, πέρα από ε, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Τράπεζα Δεδομένων, να ε, εντάσσονται σε ένα γενικότερο σύστημα όλοι οι εθνικοί λογαριασμοί και να μην είναι ε, τυχαία τα στοιχεία. Αυτοί οι συνολικοί λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν υψηλή ποιότητα, μεγάλη διαφάνεια και τα κράτη-μέλη ε, να ε, διαβιβάζουν τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορούμε σωστά να αναλύουμε την οικονομική κατάσταση σε κάθε χώρα το χρειάζονται αυτό και οι πολίτε και η τοπική αυτοδιοίκηση, δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες, διότι τα δύο τρίτα των συνολικών επενδύσεων γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Δυστυχώς όμως το σύστημα αυτό δεν είναι ακόμα πλήρε και σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2 ή ΝΑΤΣ 3 δεν έχουμε τα στατιστικά στοιχεία. Γενικά η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, προοδευτική, ε, αξιόπιστη και γι' αυτό θα υπερψηφίσω την έκθεση και παρακαλώ να πράξετε και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Τούν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αύριο θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση που μιλάει για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών. Η οι βασικέ αρχέ εκπονήθηκαν πριν από 17 χώρε, πριν από 17 χρόνια που κατάστησαν πολύ διαφορετική. Είχαμε ε, το, ε, δημιουργήθηκε τώρα η ανάγκη να ανταποκριθούμε στι νέε εξελίξει, να ενημερώσουμε τι στατιστικέ μα στην πραγματικότητα και να δούμε πώ θα διαμορφώσουμε σωστά τι ε, ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Γι' αυτό και το σύστημά μα θα πρέπει να είναι έγκαιρο, εμπρόθεσμο και ακριβές. Είναι σωστό αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τη διαφάνεια. Στην περίπτωση αυτή περιγράφουμε το δημόσιο τομέα και ο πολίτης είναι ο βασικός ε, ε, ωφελούμενος από αυτές τις διατάξεις γιατί θα λάβει πολύ πιο ακριβείς ε, πληροφορίες για την οικονομία και για την περιφερειά του και αυτό θα αποφεληθούν και οι, χώρες και οι διοικητικές αρχές γιατί στηρίζουν τις αποφάσεις μερικές φορές ε, στα στατιστικά στοιχεία. Θα πρέπει να, τηρήσουμε, να υποστηρίξουμε επίσης την ανάπτυξη των μεθοδολογιών γιατί βρισκόμαστε ακόμη στη κρίση, όλο γι' αυτό μιλάμε και η κρίση μας έδειξε πόσο σημαντική είναι η σωστή αντίληψη της κατάστασης για να προγραμματίσουμε και το μέλλον μας. Θέλουμε συνεκτικά, ενιαία και αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία για να διαμορφώσουμε σωστή αντίληψη της οικονομικής πραγματικότητας. Αυτά τα στοιχεία περιγράφουν όχι μόνο την προηγούμενη κατάσταση, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη σωστών και μεστών πολιτικών αποφάσεων και για το μέλλον, γιατί χωρίς κάτι τέτοιο η πολιτική θα είναι απομακρυσμένη από την πραγματικότητα ε, που κανονικά θα πρέπει να επηρεάσει. Γι' αυτό είμαι υπέρ αυτή τη πολύ σημαντική έκθεση για την εμπρόθεσμη και ακριβή χορήγηση πληροφοριών στατιστικών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και του λοιπού ομιλητέ και θα περάσουμε τώρα στο Catch the Eye. Δεν ήταν πολλοί που απέσπισαν την προσοχή του Προέδρου για να λάβουν μέρος στο Catch the Eye. Μόνο δύο. Ένα λεπτό έχει ο καθένας η αγαπητή κυρία Άννα Ζαμπόσκα πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει μια πιο ενδελεχής εξέταση και μέθοδος εξέτασης οικονομικής ευμάρειας και πλούτου. Γιατί η χρήση μονάχα του ΑΕΠ οδηγεί σε στρεβλώσεις το ΑΕΠ να αντανακλά το έργο των νοικοκυριών που λαμβάνει χώρα στα νοικοκυριά. Ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι στα νοικοκυριά δεν αντανακλάται στο ΑΕΠ. Και φυσικά παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας και υποτιμάται ο ρόλος των γυναικών και η εργασία των γυναικών. Αν λοιπόν με τον τρόπο αυτό μειώνουμε το χρόνο που δαπανούν οι γυναίκες για να φροντίσουν τα παιδιά τους, αυτό δεν αυξάνει την ευμάρεια. Εμείς απλώς θεωρούμε ότι είναι θετικό να πληρώνει η μητέρα κάποιον να φροντίζει τα παιδιά τους αντί να τα φροντίσει η ίδια. Ευχαριστώ Άννα. Και ο Λουκούμιος, ο μιλητής, για ένα λεπτό είναι ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παροχή και η διαβίβαση στοιχείων για τους λογαριασμούς των κρατών μελών είναι προαπαιτούμενο για να μπορούμε να καθορίσουμε σωστά τις οικονομικές πολιτικές. Η βελτίωση των οικονομικών συστημάτων για τους εθνικούς και περιφερειακούς λογαριασμούς θα πρέπει επομένως να συμβάλλουν στο να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για να μπορούν να αντανακλούνται οι πραγματικέ οικονομικέ συνθήκε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλύτερη αξιολόγηση με ρεαλιστικό τρόπο των οικονομικών συνθηκών. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν αξιόπιστα στοιχεία τα οποία να μπορούν να έχουν μια ενιαία μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε αυτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την αίτηση της έκθεσης που ζητά από την Κομισιόν να το τροποποιήσει το σύστημα για την παροχή και συλλογή στοιχείων στην περίπτωση που δεν είναι πλήρη τα στοιχεία αυτά, δεν είναι απλά και δεν είναι και διάφανα. Σας ευχαριστώ, λέει ο αγαπητέ συνάδελφε. Τελείωσε και αυτή η διαδικασία. Και για να κλείσουμε τη συζήτηση θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Ποτότσνικ, εξ ονόματος Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κάποιες επεξηγήσεις ίσως γιατί όπως αναφέρθηκε υπάρχει το θέμα των ε, δυνητικών ε, στοιχείων ε, παθητικού σε επίπεδο των εθνικών λογαριασμών. Το θέμα αυτό παρουσιάστηκε στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, η οποία έδωσε την υποστήριξή της και η συλλογή αυτών των στοιχείων για τα χρέη των ε, συμπράξεων ιδιωτικού και θετικού και δημοσίου τομέα και ιδιωτικού και επίσης τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος θα οδηγήσουν σε εκθέσεις που θα είναι διαθέσιμε το 2014 για τις συντάξεις θα, θα δίδονται από το 2015 υποχρεωτικά σε τριετή βάση και τέλος η Κομισιόν είναι έτοιμη να παρουσιάσει μια έκθεση προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, μάλλον η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, την ΕΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν το ζητήσει. Είπατε ότι είναι βαρετό αυτό το θέμα. Για πολλά χρόνια εγώ ήμουνα επικεφαλής μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Στατιστικής Οργάνωσης στη Σλοβενία και έχω πάρει και διδακτορικό για τα θέματα των εθνικών λογαριασμών και ξέρω περισσότερο για το S95 από ότι οποιοδήποτε άλλο εδώ κατά πάσα πιθανότητα. Μπορώ να σας πω ότι καμία από τις σημαντικές και ουσιαστικές αποφάσεις δεν μπορεί να λαμβάνεται χωρίς εργόδη στατιστική επεξεργασία και οι μακρές μεθοδολογικές συζητήσεις είναι και αυτές απαραίτητες και είδα ότι η η ΕΣΑ είναι μια στατιστική βίβλος για όλους μας. Με το να την ενημερώσουμε από το 95 στο τωρινό σύστημα, εξασφαλίζουμε σταθερότητα στο στατιστικό σύστημα και προσθέτουμε νέα στοιχεία που αντανακλούν τη νέα γνώση και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσει. Μπορεί να φαίνονται ανιαρά όλα αυτά, αλλά χωρίς σκληρή εργασία δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να παίρνουμε σημαντικέ και δίκαιε αποφάσει. Σα ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω από την πλευρά τη Κομισιόν στο να συνεχίσουμε αυτό το έργο και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση με την παρέμβαση της αγαπητής κυρίας Μπόουλς ε, της εισηγήτριας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν σας αρέσει η αιτιολογική σκέψη 16, αλλά τα οικονομικά θέματα είναι ε, εξαιρετικά και έκτακτα αυτές τις περιστάσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι από τους πρώτους χρήστες και θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο να μπει ε, και να έχει δικαίωμα διαβούλευση και για τις ε, κατεξουδότηση πράξεις ε, έχουν αυτό το δικαίωμα για όλες τις πράξεις και το θεωρούσαμε κατ' επέκταση δικαίωμά τους. Και εσείς και η κυρία Φόρτ και ο κύριος Γκίγκολτ αναφερθήκατε στο θέμα των στοιχείων παθητικού, θα επανέλθω στη συνέχεια ε, σύντομα. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική διαβίβαση έχουμε βάλει ασφαλιστικές δικτυλίδες περισσότερες και μεταξύ αυτών ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αναφέρει για οποιαδήποτε στοιχεία έχει για τις ΔΙΤ και άλλες ε, έμεσες ε, ή ε, όχι ε, πρόδειλες περιπτώσεις στοιχείων παθητικού. Θα το παρακολουθούμε αυτό πολύ στενά και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και δείχνει ότι έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν μπορούμε 15 χρόνια ε, να έχουμε στοιχεία από το 1995 ε, και συστήμα θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα και εργαζόμαστε ήδη για το επόμενο θέμα των στατιστικών που έχει να κάνει με τη λειτουργία του στατιστικού πλαισίου και την εξαρτησία των στατιστικών αρχών. Είναι ο κανονισμός 223 όπως είναι γνωστό στη γλώσσα μας. Ε, δυστυχώς μέχρι τώρα τι ακούω ότι τα κράτη-μέλη και πάλι να πρόκειται πρόθυμα να υπογράψουν για να μην μπορούν να συζητήσουν καν αυξημένη διαφάνεια. Δηλαδή στην ιστοσελίδα τους να δια, βιβάζουν και να δημοσιεύουν τις υποχρεώσεις αυτές στα κράτη-μέλη. Περίεργα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ε, έρχομαι στο θέμα του ΕΣΑ 2010 ε, και παρακαλώ να υπερψηφίσετε την έκθεσή μου και με την υποστήριξη της Επιτροπής θέλουμε να κλείσει σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ κυρία Μπόουλς. Με τη δική σας παρέμβαση ως ηγήτρια τελειώνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει όντως αύριο. Αύριο το μεσημέρι στις 12. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη η απόψε είναι η έκθεση της κυρίας Βέσλουντ με θέμα την προστασία της δημόσιας υγείας από ουσίες που